Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Καθίστε παρακαλώ. Και παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση κατευθείαν με το σημείο 12 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημείο 12. Αλλά παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ζητήσω από την κυρία Ματέρα, την εισηγήτρια, να μας πει αν θέλει το λόγο. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Αρχίζουμε τη συμβαστική ψηφοφορία 1. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ σηκώστε το χέρι. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά,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 Απολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβεστική 3 υπέρ Συγγνώμη, συγγνώμη. 18 έγινε δεκτή, τότε καταπίπτει η συμβαστική. Περνάμε στην 21, τροπολογία 21. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 23. ψήφι, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε πύρις 23 πέρας της το ΕΛΚ ε, έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι δικαιούται όχι τώρα εντάξει, εντάξει απορρίπτεται η τροπολογία Τροπολογία 24 πρόκειται για χωριστή ψηφοφορία. Όχι, όχι, δεν είναι χωριστή ψηφοφορία, αν κάνω λάθος. Ψηφίζουμε επί της 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 καταπίπτει. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ψηφίζουμε επί της 25. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 36 υπέρ 36 ναι. ψηφίζουμε επί της 36 Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν κοιμηθεί καλά απόψε. Τροπολογία 34. Ψηφίζουμε επί 34. Ψήφι υπέρ. <coughs> Κατά. Αποχές. Ας γίνει επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί τη 34. Δεκτή. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου δεν ακούστηκε. Υπάρχει μία ψήφος του ΕΛΚ περισσότερη από ό,τι δικαιούστε. Δεν είναι δική μου, είμαι πλήρες μέλος. Αν θέλετε, παραλάβαν με την ψηφοφορία, αλλά κάποιος από το ΕΛΚ θα πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα του. Ξαναψηφίσουμε επιστροπολογίες 34, άρα για την ψηφοφορία. 26 μέλη θα πρέπει, θα πρέπει να είναι παρόντα. Ακόμα ένας πρέπει να βγάλει την κάρτα. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως έχει εγκριθεί αλλά σε ελέγξουμε καλού κακού 39 τροπολογία άρχιτη ψηφοφορία επί της 39 Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση επί τη 41. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 41. Πέρα ψηφοφορίας έγινε δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Και εγώ καταψήφισα. Παρατηρεί κάποιος, κάποιος από την αίθουσα, εκτός μικροφώνου. Αλλά υπάρχει ένα άτομο παραπάνω από το έλκυο. Αποφασίστε ποιος θα πρωτοψηφίσει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δικαιούστε πάνω από 12 ψήφους. Κοιτάξτε, ένας από το ΕΛΚ θα πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα από το μηχανάκι. Εντάξει, θα επαναλάβω την ψηφοφορία. Εντάξει, σας υπόσχομαι θα κερδίσετε, αλλά τόση μην ψηφίζετε παραπάνω άτομα. Λοιπόν, ψηφίζουμε εκ νέου επί της 41. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 41. Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία. 42. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα η ψηφοφορία στην Λίμπε θα γίνει στις 19 ε, Ιουνίου. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, παρελθόν 13, εφαρμογή της Ραγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία 2010-2012. Ο εισηγητής, θα επιθυμεί να λάβει το λόγο. Τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Δεν θα τις ψηφίσουμε ομού, αλλά μία προς μία. Ξεκινάμε με την υπαριθμόν 5 ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα περνάμε στο σημείο 14 για τον προγραμματισμό πολιτική και μακροπρόθεσμη στάση στι δημοσιονομικέ επιπτώσει τη δημιουργία ικανοτήτων. Μπορούμε να ψηφίσουμε ομού όλε τι Μάλιστα, άρα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Περνάμε στο σημείο 15 καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Κάνω κάποιες ανακοινώσεις επί της 81 και 82. Ε, αναφέρεται το όνομα του συναδέλφου Σκούρια Μάλλον δεν αναφέρεται και το, το καταγράφουμε όμως, έγιναν κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά θέματα της χωριστή ψηφοφορίας. Ίσως η κυρία Αντζελίλη θα θέλει να μας εξηγήσει το ζήτημα αυτό. Συγγνώμη, κυρία Αντζελίλη, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τροπολογία 79 Νομίζω πως ε, περιέχει κάποιο σφάλμα. Έχει ζητηθεί λοιπόν χωριστή ψηφοφορία το πρώτο τμήμα που ξεκινάει με το ότι δημιουργεί τα κράτη-μέλη και καταλήγει εισόδημα των γυναικών ε, σε σχέση με το εισόδημα των ανδρών και δεύτερο τμήμα τονίζει την ανάγκη για την εφαρμογή και καταλήγει με το ε, και οι γυναίκες και οι άντρες. Both women and men. Αυτή είναι μια τεχνική τύπου διευκρίνηση που θα θέλω να κάνω. Ε, όπως είπε η κυρία Αντζελίλη, η πρόταση που λέει stresses, the need to implement, INCO ε, κλπ. Δεν θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι της πρώτης χωριστή ψηφοφορίας. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο δεύτερο κομμάτι της ε, τροπολογίας ε, Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβαστική 6 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβαστική 9 υπερ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 36 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση επί τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία με τη 42. Απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Προπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα επαληθεύσουμε για τη 46. Άρχεται ψηφοφορία για τη 46. Ε, πέρα ψηφοφορίας έχει απορριφθεί η τροπολογία. 47 ψήφι υπέρ. Κατά εποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε για την 62 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας ε, εγκρίθηκε. 56 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 66. Εγκρίθηκε μία ψήφο διαφορά. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συνδεστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συνδεστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 78. πέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίθηκε. Χωριστή ψηφοφορία επί της 79. Α μίλησε κυρία Αντζελίλη για αυτήν. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, εποχές. Ας επαληθεύσουμε καλού κακού, πρώτο τμήμα τη τροπολογίας 79, τροπολογία 79, πρώτο κομμάτι αυτή. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας, ψηφιπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 81, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 85, 87 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε γιατί δεν ψήφισαν δεν σήκωσαν τα χέρια του Άρχιε ψηφορία για την 87. Πέρα της ψηφορίας. Απορρίφθηκε. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συνδεστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας απελθεύσουμε λοιπόν για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τοπολογίας 25. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορριφθήκε. 27 υπέρ. Κατά. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 28 έχει υποσυρθεί. Περνάμε στην 29 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επί του συνόλου ψηφίσματος. Ναι, παρακαλώ κυρία Αντζελίλη, έχει το λόγο. Πρόεδρε πριν προσπάθησα να σας κάνω νόημα για να σας πω ότι ήθελα έλεγχο για την τροπολογία 81. Συγγνώμη, πήγαμε γρήγορα, προχωρήσαμε, προσπάθησα να σας το υποδείξω, αλλά δεν με είδατε. Ωραία, για μια ακόμα φορά λυπάμαι για το συμβάν. Κύριε Αντζελίλη, φυσικά μπορείτε να, να κάνετε νοήματα και να κραυγάσετε, αν θέλετε να την προσοχή μου. Περνάμε λοιπόν στην 81 εκ νέου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 81. άρχιτη ψηφοφορία επί της 81. Πέρα ψηφοφορίας έγινε δεκτή. Τώρα επί του συνόλου του ψηφίσματος, άρχιτε ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε ξεκάθαρα το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σημείο 16. 16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 κατά αποχές εγκρίνεται ε, ας επαληθεύσουμε για τη 16 άρχεται ψηφορία πέρας εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 έχει 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία Α, να επαληθεύσουμε για την 21, ωραία. Επαλήθευση της 21 άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία και θα ζητήσω αν υπάρχουν ενστάσεις επί της προφορικής τροπολογίας. Όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Επαλήθευση επί της προφορικής τροπολογίας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί του συνόλου του ψηφίσματος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Έγινε δεκτή. Συγχαρητήρια στην συγκεντρία. Περνάμε στι διασυνοριακέ συλλογικέ διαπραγματεύσει και τον διεθνικό κοινωνικό διάλογο. Ξεκινάμε με τον συμβασμό 1, ψηφιπέ, κατά αποχές δεκτή την τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12, χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα με υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές Επαλήθευση επί της 14 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας έγινε δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή καταπίπτει 18, περνάμε στην τροπολογία 19, ψηφιπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24 καταπίπτει, περνάμε στην 25, ψηφιπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 καταπίπτει 34 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές ευρύνεται 36 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 37 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, Τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε επί τη 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. απορρίφθηκε. Τοπολογία 3 υπέρ κατά αποχές ε, Δύο χωρίς την ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πρώτο για τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεργαστική 3 υπέρ κατά εποχές ε, εγκρίνεται, τροπολογία 6 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται, τροπολογία 7 έχει καταθέσει, τροπολογία 8 επίσης, ψηφίζουμε επί του συνόλου του ψηφίσματος, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Σαφές το αποτέλεσμα, έγινε δεκτή η έκθεση. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία, υπερθυμών 18 και ξεκινάμε με την τροπολογία 20. Ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ψηφίζουμε για την προπολογή 25 Έληξη ψηφοφορία έγινε δεκτή. Προπολογία 23, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά πρέπει να επαληθεύσουμε ψηφίζουμε επί 26 26 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση επί της 29 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 31 έχει αποσυρθεί 31 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 33 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ, κατά αποχές δεκτή επαλήθευση επί τη 42 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε Προπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα επαληθεύσουμε επί τη 40 άρχιτη ψηφοφορία ε, πέρα ψηφοφορίας και έχει απορριφθεί 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος επί της 3 ξέρετε η υποψηφία αλλάζει κάθε φορά τροπολογία 3 λοιπόν άρχισε η συγχωρία Έληξε η ψηφοφορία και έχει εγκριθεί. Προπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, επαλήθευση. Προπολογία 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ναι, ναι. Είχε απορρευθεί. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση επί της συμβαστικής 2. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 και 16 δεν ε, ψηφίζουμε πέραν 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές ε, συγγνώμη 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος άρχιτη ψηφοφορία ηλεκτρονικός Πέρα της ψηφοφορίας, σαφής η έγινε δεκτή ε, η έκθεση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την, ε, την συντάκτρια. Να σας πω ότι η ψηφοφορία μου ήταν θετική, διότι το μηχάνημά μου μπλοκάρισε. Υπερψήφισα λοιπόν.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 Då återupptar vi de här förhandlingarna och nu så är, pratar jag... Om jag då I'm not going speak Swedish uh, because I'm gonna open up the meeting. Θα μιλήσω σουηδικά. Και θα ξεκινήσω με κάποια ε, σημεία διοικητικά πριν περάσουμε στη φιλοξενούμενη. Θα, θα μιλήσω σου ειδικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν την συνεδρίασή μας. Έχουμε κρίνει την ε, ημερήσια διάταξη, τη στιγμή δηλαδή που δεν υπήρξαν κάποιες ε, άλλες ε, απόψεις. Έχω κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να κάνω τις ανακοινώσεις μου. Πρώτον, θα γίνει μια συνάντηση με κυρία Βαμπαγκούρα για μεσημεριανό εκπρόσωπο για θέματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλικά προβλήματα. Αυτό θα γίνει ανάμεσα στη 1.30 και στις δύο. και το απόγευμα επίσης θα έχουμε μια ακρόαση η οποία αφορά δράσεις. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. λοιπόν, 20 Ιουνίου θα έχουμε μια ακρόαση. Το απόγευμα θα έχουμε μια άλλη ακρόαση για γυναίκες με ειδικέ ανάγκες. Αλλά μετά θα έχουμε την ακρόαση για θέματα που έχουν να κάνουν με τις ε, εκλογές και με την ισορροπία ανάμεσα ε, ε, στα δύο φύλλα. Αυτά 20, 20 Ιουνίου. Τώρα, επίσης ενημέρωση για τις δράσεις των που έχουν γίνει. Έχετε λάβει κάποια έγγραφα. Αν δεν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Επίσης, Επίση στο σημείο 5 έχω το θέμα των πρωτοκόλων μια σειρά συναντήσεων, τα πρακτικά δηλαδή. Επίση, έχουμε τα υπόλοιπα από τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο κτλ. Και όλα αυτά τα, τα πρακτικά θα θεωρούνται ε, ότι έχουν εγκριθεί αν δεν υπάρχει κάποια, ε, κάποιο σχόλιο. Τώρα λοιπόν περνάμε στο ενδιαφέρον θέμα. Και χαίρομαι ότι δίπλα μου βρίσκεται η κυρία Τάιτεμπαουμ από το θα λέγαμε Ευρωπαϊκό Γυναικείο Λόμπι. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι όλα τα μέλη που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ασχολούνται μαζί τους, ρωτάνε, παίρνουν συμβουλές. Είναι μια οργάνωση ομπρέλα σε, για μια σειρά οργανώσεων που βρίσκονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και εκπροσωπούν επίσης και τρεις υποψήφιες χώρες. Να τη χαιρετήσω λοιπόν εδώ πέρα, χαίρομαι που την έχουμε μαζί μας, θα κάνουμε κάποια ερωτήματα, θα ανταλλάξουμε ιδέες και προβληματισμούς, αλλά καλύτερα να σου δώσω πρώτα το λόγο να κάνεις την εισαγωγή σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Good morning and... Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ, Μάικλ, κύριε Γκούσταυσον. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκλησή σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών, που παίζει σημαντικό ρόλο για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ούτως ώστε να βάλουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην πολιτική σε διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις πολιτικές. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που κάνετε και για το ενδιαφέρον σας και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στη συνεργασία με οργανισμούς ε, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Όπως ξέρετε και όπως είπε και ο κ. Γκούστευσον, το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ε, είναι ο μεγαλύτερος συνασπισμός ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και έχουμε μέλη και σε όλα τα, και εκτός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κροατία, Μακεδονία, Τουρκία και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ε, επίκαιρο το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω εκ μέρους όλων των γυναικών που εκπροσωπούμε και για να συμμεριστούμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα τελευταία πέντε χρόνια τα μέλη μας μας ενημερώνουν συνεχώς για τις επιπτώσεις καταρχήν της κρίσης και για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις ζωές των, στις ζωές των γυναικών. Βλέπουμε μια ανησυχητική τάση επανιδιωτικοποίησης της περίθαλψης που πολύ συχνά οδηγεί στο ότι οι γυναίκες ε, ε, επαναπέμπονται ε, στο σπίτι τους, εκτός νοσοκομιακών δομών δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν δομές για την περίθαλψη των παιδιών ή των ηλικιωμένων και οι γυναίκες αναγκάζονται να επιστρέψουν στην στο νοικοκυριό του. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζει λοιπόν τεράστια προβλήματα και αυτό αποτελεί και ένα κίνδυνο ένδυα ε, λόγω της διαφοράς ε, στις αμοιβέ και στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκτός από το ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών, η κρίση χρησιμοποιείται και ως πρόφαση για να φυγούν τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Οι θεσμικοί μηχανισμοί όπως οργανισμοί ισότητας ή υπουργικέ δομέ έχουν αποδυναμωθεί και δεν υπάρχει δημοκρατική ισότητα στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν όλο και περισσότερες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών ε, με τρόπο κάπως οργανωμένο. Από τη μια πλευρά ε, οι γυναίκες ε, επαναπέμπονται στον παραδοσιακό ρόλο του ότι αναλαμβάνουν να φροντίζουν τα αδύναμα μέλη και είναι ο δεύτερος παράγων στην οικογένεια όσον αφορά τη συνεισφορά στο εισόδημα και αυτό οδηγεί την διαιώνιση των στερεοτύπων του φύλου για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, όπου η προτεραιότητα δίδεται στην απασχόληση για τους άνδρες και τη γυναίκα στο σπίτι. Αυτό έχει επιπτώσεις και στις επιλογές που κάνουν τα κορίτσια όσον αφορά την παιδεία και την σταδιοδρομία τους και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει υπερσεξουαλικοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και γίνεται εμπορευματοποίηση της διαφήμισης και εκπορνισμός του δημοσίου χώρου. Βλέπουμε όλο και περισσότερες εικόνες που μεταφέρουν το μήνυμα ότι τα σώματα των γυναικών και η σεξουαλικότητα των γυναικών προσφέρονται για τις φαντασιώσεις των ανδρών και προωθούνται προωθείται η εμφάνιση περισσότερο έναντι της αυτοεκτίμησης των γυναικών. Υπάρχει άμεση επίπτωση λοιπόν στις σχέσεις ανδρών και γυναικών και στο πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια στη βία των ανδρών. Αυτές οι τάσεις λοιπόν έχουν τους ίδιους στόχους, έλεγχο του σώματος και της σεξουαλικότητας των γυναικών και περιορισμό της ελευθερία των ε, γυναικών. Χαίρομαι που η Επιτροπή για τα Δικαιώματα τη Γυναίκα ε, θα συζητήσει βασικά ζητήματα τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα πέραν της δουλειάς σας ε, για τα ε, τρία θέματα, βία κατά των γυναικών, σεξουαλικά δικαιώματα και πορνεία, θα επανελάβουν ε, το ισχυρό φεμινιστικό μήνυμα ότι οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γκούστασον ότι έχουμε τους ίδιους στόχους. Θέλουμε οι γυναίκες και τα κορίτσια να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς παρεμβάσεις στις επιλογές τους, ούτε θρησκευτικέ, ούτε πολιτικές, ούτε κοινωνικές, ούτε οικονομικές. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές ε, τις, αυτούς τους συσχετισμούς μεταξύ υπερσεξουαλικοποίησης και βίας κατά των γυναικών. Θα ήθελα να πω δύο λόγια τώρα και για τα σεξουαλικά δικαιώματα και την πορνεία προσπαθώντας ε, να σας τροφοδοτήσω με κάποια θέματα προς συζήτηση και σκέψη. Το θέμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων είναι κυρίως θέμα δικαιωμάτων των γυναικών και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των ε, διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών βλέπουμε ότι υπάρχει μια οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην Ευρώπη και νέες στρατηγικές να εμποδίσουν την πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη για την αναπαραγωγική υγεία. Έχουν μειωθεί ε, λόγω των μέτρων λιτότητας έχουν μειωθεί οι υπηρεσίες υγείας για τη σεξουαλική και ε, αναπαραγωγική υγεία και στην Γαλλία, παραδείγματος χάρη, 180 κέντρα αμβλώσεων αναγκάστηκαν να κλείσουν τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης βλέπουμε αυξανόμενη πίεση θρησκευτικών ομάδων κατά της αυτοδιάθεσης των γυναικών όσον αφορά την αναπαραγωγική τους υγεία. Το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη, οι τρέχουσε συζητήσεις σχετικά με την άμβλωση στην Ισπανία και στην Ιρλανδία ε, όπως επίσης ε, και η χρήση των ε, Τη αντίρρηση συνειδήσεως που εμποδίζει τις γυναίκες από την πρόσβαση σε υπηρεσίες αμβλώσεων ακόμη και σε χώρες όπου η άμβλωση είναι νόμιμη. Εκτός από την άμβλωση υπάρχουν και επιθέσεις σε ολόκληρο το φάσμα των δικαιωμάτων των γυναικών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, αντίδραση στην ε, ε, κοινή εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών σε πολλές χώρες, κυρίως υποκινούμενοι από θρησκευτικέ ομάδες, παρά την έκθεση του ειδικού ε, του των Ηνωμένων Εθνών το 2010 σχετικά με το δικαίωμα για την εκπαίδευση που ε, διακηρύσει ότι ε, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και το δικαίωμα σε ε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για την δυνατότητα μεθόδων αντισύλληψης και πολλές γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στα αντισυλληπτικά διότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρά. Επίσης υπάρχει το θέμα των γυναικών που χρησιμεύουν ως υποκατάστατο μητέρας για, μητέρες που δεν μπορούν να για γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν γεννήσουν παιδιά ε, και θα θέλαμε επίσης ε, να επιστήσουμε την προσοχή ε, στο πόσο, πόσες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό στα σεξουαλικά δικαιώματα της γυναίκας και στην εμπορευματοποίηση του σώματος των γυναικών. Επίσης συνεχώς θα πρέπει να παραπέμπουμε στις επιπτώσεις της βίας των ανδρών στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Πολύ σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε και τις ειδικέ ανάγκες των γυναικών. Οι γυναίκες Ρωμά και οι γυναίκες με αναπηρία στην Ευρώπη άνθρωποι ε, συχνά αντιμετωπίζουν επιβεβλημένη στήρωση που αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ακαιρεότητας ε, ε, του σώματος των γυναικών, την ελευθερία επιλογής τους και το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση και αναπαραγωγική υγεία. Άλλο ένα θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι η πορνεία, η σεξουαλική εκμετάλλευση και η επίπτωση στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη. Τονίζω λοιπόν την ανάγκη να επανέλθουμε στο ευρύτερο πλαίσιο των διαθροτικών ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ελπίζω πραγματικά ότι η δουλειά σας για τα θέματα αυτά θα ξεκινήσει αναγνωρίζοντας το ότι έχει σχέση με το φύλλο, το φαινόμενο της πορνείας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δεν μας εκπλήσει που η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εκπορνευωμένων προσώπων είναι γυναίκες και η πλειοψηφία των αγοραστών σεξ είναι άνδρες. Και βεβαίως αυτό έχει σχέση με τις πατριαρχικές δομές της κοινωνίας μας και με στερεότυπα σε σχέση με το φύλλο και την ε, αιμονή της ηγεμονικής ε, θέσης των ανδρών που ε, δικαιολογεί το να διατίθενται ορισμένες γυναίκες για τις αποκαλούμενες ανάγκες των ανδρών. Χρησιμοποιώ τη λέξη σύστημα, διότι υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που εμπλέκονται στο θέμα της πορνείας και πρέπει να εξετάσουμε τους ρόλους όλων αυτών όταν αντιμετωπίζουμε την επίπτωση της πορνείας στην ισότητα των φύλων. Το σύστημα της πορνείας ε, πηγαίνει πιο μακριά από το παραδοσιακό θέμα των ατόμων που εμπλέκονται στην πορνεία. Περιλαμβάνει και τους αγοραστές. Και είναι σαφές ότι χωρίς τους αγοραστές δεν θα μπορούσε να υπάρχει πορνεία. Αυτοί αποτελούν τη ζήτηση που τροφοδοτεί την ε, προσφορά και η πορνεία έχει επιπτώσεις και στους άνδρες. Το σύστημα της πορνείας συμπεριλαμβάνει επίσης ε, και τους προαγωγούς, ε, τους προμηθευτές και τους εμπόρους ε, ανθρώπων που εποφελούνται οικονομικά από την πορνεία άλλων. Οργανώνουν ολόκληρο αυτό το σύστημα πορνείας, το έχουν μετατρέψει σε μια βιομηχανία σεξ και χρησιμοποιούν την παγκοσμικοποίηση για να εκμεταλλευτούν τους πλέον ευάλωτους. Τα εκπονευόμενα πρόσωπα είναι στην ε, πλειοψηφία τους γυναίκες και κυρίως γυναίκες από τρίτες χώρες ή από μειοψηφίε ή από ομάδες ε, που αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Άμστερνταμ και στη Ζηρίχη οι γυναίκες Ρωμά ε, αντιπροσωπεύουν το 80 έως 99% των εκπορνευόμενων γυναικών που προέρχονται από την Ουγγαρία. Το σύστημα της πορνείας συμπεριλαμβάνει και την κοινωνία επίσης, δηλαδή εμάς, τους πολίτες και τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τους λαμβάνοντες αποφάσεις, εσάς δηλαδή όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε γιατί οι πολιτικές μας μπορούν είτε να υποστηρίξουν το σύστημα της πορνείας είτε να το καταγγείλουν και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι πολιτικές επιλογές μας έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες στα άτομα που εμπλέκονται στο σύστημα της πορνείας και γενικότερα σε όλους μας στις απόψεις της κοινωνίας για τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και στις, ε, στην εντύπωση που έχουν οι νέοι για ε, την σεξουαλικότητα και την ισότητα. Ελπίζω λοιπόν ότι η δουλειά που κάνετε για αυτά τα θέματα θα αντιμετωπίσει όλους τους παράγοντες του συστήματος και θα ακολουθήσει μια πραγματική ανάλυση του τι σημαίνουμε τι σημαίνει η ισότητα των φύλων και όταν αντιμετωπίζουμε το θέμα της πορνείας και τι θέλουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έχει μια ισχυρή θέση στο θέμα της πορνείας από το 1998. Εμείς τονίζουμε ότι η πορνεία σαφώς αποτελεί καταστρατήγηση των, δικαιω... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Και χαιρετίζω την τελευταία έκθεση ε, της Επιτροπής ε, Γυναικών ε, που κατατάσσει την πορνεία μεταξύ των μορφών βία κατά των γυναικών. Και αυτό αποτελεί επίτευγμα τη επιτροπή σα. Πιστεύουμε ότι η πράξη τη πορνείας που αποτελεί μια σεξουαλική πράξη η οποία διαπράτεται χωρί επιθυμία και ε, λόγω ανάγκη για χρήματα είναι επιβλαβή για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ατόμου. Όπω γνωρίζετε υπάρχει βία στην πορνεία. Σπανίως μιλάμε για την επίπτωση της πορνείας ε, στην ψυχική και σεξουαλική υγεία των εκπορνευομένων προσώπων ή στην ευημερία τους και στην αυτοεκτίμησή τους. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με το χώρο, η βία του συστήματος της πορνείας έγινε στην πραγματικότητα ε, την οποία τα εκπρονευόμενα άτομα αναγκάζονται να συνενέσουν στην παραβίαση της αξιοπρέπειάς τους αποδεχόμενα μια σεξουαλική πράξη σε μια μη ίση κατάσταση. Αν υπήρχε ισότητα δεν θα υπήρχε ανταλλαγή χρημάτων. Όπως λέει κάποιος ε, στην, ε, στο ντοκιμαντέρ Not for Sale, δεν ε, πωλείται, αν οι γυναίκες είχαν περισσότερες επιλογές όσον αφορά την οικονομική τους συμμετοχή σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα επέλεγαν να είναι αντικείμενα εκμετάλλευση στην πορνεία. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν εδώ τις πραγματικές ρίζες, τις πραγματικές αιτίες και τις επιπτώσεις της πορνείας στην ισότητα των φύλων και ελπίζω ότι θα λάβετε υπόψη τις φωνές των επιζώντων, γιατί πραγματικά επιζώντες είναι αυτοί που επιβιώνουν από το δίκτυο της πορνείας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά πώς θεωρούμε εμείς το ρόλο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος για την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε στη δουλειά σας και στις προσπάθειές σας να εντάξετε την πολιτική των φύλων σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι θα αναπτύσσετε τα περισσότερες στρατηγικές στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει ένα πιο ισχυρό ρόλο και θα εντείνει το διάλογο μεταξύ των, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουμε προοδευτικές πολιτικές ε, για να αλλάξουν οι ζωές των πολιτών με θετικό τρόπο. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών σήμερα στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για αυτήν εδώ την εισαγωγή και όπως είπες ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτά τα μηνύματα που μας δίνεται και συμφωνώ μαζί σου ότι ε, ε, χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας και εδώ στην Επιτροπή μας συζητήσαμε διάφορες εκθέσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα όσον αφορά τη σεξουαλική διάσταση. Ε, εγώ προσωπικά ε, ε, έχω ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα το οποίο ακριβώς έχει να κάνει με τον τρόπο που οι άντρε εκμεταλλεύονται το γυναικείο κορμί. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσά μας ούτως ώστε ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να λάβουν ε, γνώση για την εμπειρία σας και να δούνε τι ακριβώς γίνεται γύρω στον κόσμο. Τώρα θα δώσω τη δυνατότητα στα μέλη να κάνουν ερωτήσεις αλλά πριν θα ήθελα να πω. Έχουμε δύο ομάδες επισκεπτών. Η μία ομάδα από τη Μωρή Σαρτιέ έχει ε, κληθεί εδώ και τους καλωσορίζουμε. Και, ε, έχουμε μια άλλη ομάδα που έχει να κάνει με μελέτες για τα γυναικεία θέματα και χαιρόμαστε που τους έχουμε και αυτούς εδώ, αυτές μάλλον, ε, ε, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι τι, πιστεύετε, ποια εντύπωση δημιουργείται μετά από αυτήν εδώ την επίσκεψη. Λοιπόν, ξεκινάμε ε, με την Μωρίν ε, Σαρτιέ πρώτη-πρώτη, η οποία θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία ε, Τάιτελμπάουμ που είναι μαζί μας σαν αντιπρόεδρος που είναι του Ευρωπαϊκού Λόγου Γυναικών. Χαιρετίζω φυσικά αυτήν εδώ την επίσκεψη και είναι σημαντικό να υπάρχει κινητοποίηση. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο, το πρώτο που θίξατε. Η επιπτώσεις της κρίσεως στις γυναίκες και κυρίως την ε, εργασία των γυναικών. Θα ήθελα και η μεν και η δε των διαφόρων, τα διάφορα, στα διάφορα δίκτυα να είναι πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό το θέμα διότι κατ' εμέ η εργασία είναι το βασικό μέσο για την ανεξαρτησία των γυναικών και για την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Αλλά με την κρίση τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι πρώτον οι γυναίκες σφαιρικά αν το δούμε έχουν ένα μισό ο οποίος είναι ευρέως ε, πολύ χαμηλότερος από αυτό τον των ανδρών και σοκάρει αυτό. Ε, και όλα αυτά εν ονόματι της ισότητας των πολιτών. Θα πρέπει όντως να κινητοποιηθείτε και εμείς θα το κάνουμε πολιτικά από τη δική μας πλευρά. Ε, λοιπόν, ισότητα μισολογική. Δεύτερον, τα θέματα της ισότητας όσον αφορά τον διάφορους τύπους συμβόλων στις γυναίκες και στους άνδρες. Τι βλέπουν, πολλές γυναίκες έχουν ε, ε, επισφαλή απασχόληση ε, και υπερέχουν σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδιο και στην μερική απασχόληση. Αυτά δηλαδή βλέπουμε έχουν επιδονθεί στα πλαίσια της κρίσης. Και είναι αυτά που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτή η μερική απασχόληση Φερρυπίν ε, οδηγεί σε μια κατάσταση όπου είναι και τα, οι πρώτε θέσει που πλήττονται και καταργούνται σε σχέση με την κρίση. Τώρα, αν προσθέσετε τώρα, χαμηλή μισολογία, μερική απασχόληση, δυσκολίες καθημερινές, συνδυασμός εκεί προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, βλέπουμε οι γυναίκες έχουν υποχωρήσει σιωπηλά από το χώρο της εργασίας. Απ' τη μια θέλουμε κινητοποίηση για να εξασφαλίσουμε την ισότητα άνδρες γυναίκες στην καριέρα, μισολογία, στη, στη θέση που έχουν, αλλά ταυτόχρονα και γι' αυτό απευθύνουμε τώρα σε εσά να κινητοποιηθούν οι γυναίκες ούτως ώστε πραγματικά να παλέψουν, να αντισταθούν να έχουν ίση αμοιβή και ίση θέση με σχέση με τους άνδρες. Αν δεν το κάνουμε μαζί από κοινού, στο τέλος της επαγγελματική ζωής τι διαπιστώνουμε, οι γυναίκες περνάνε στην, ε, στην ε, σύνταξη με 33% λιγότερη αμοιβή από τους άνδρες. Και έχουμε την φτώχεια των γυναικών και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί ενισχύεται σήμερα η φτώχεια των γυναικών και μελλοντικά πολιτικά θα αποτελήσει οικονομικό και κοινωνικό μεγάλο πρόβλημα. Κινητοποίηση λοιπόν ξανά. Γι' αυτό το λέγω σε σχέση με την έκθεση που έκανα εγώ για την επιπτώση της κρίσης στην εργασία των γυναικών ε, έκανα τα πάντα και ελπίζω όλοι μαζί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν μια έμφαση και δεν είναι μόνο ο συνδυασμό ε, επαγγελματικής και οικογενειακή ζωής για την γυναίκε, αλλά και το θέμα της γυναικείας καριέρας. Με. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη θα πάρει το, το λόγο. Thank you very much. Ε, I... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η νέα τάση ότι οι άνδρες πρόσφατα συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και της αξιοπρέπειας των γυναικών. Ξεκίνησε και από τον τομέα της πατρότητας και σιγά σιγά οι άνδρες συνόδευαν τις γυναίκες τους κατά τη διάρκεια του τοκετού και περνούσαν όλο και περισσότερο χρόνο με τις συζύγους και το παιδί. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούσαν οι πατέρες να συνδεθούν καλύτερα με τα παιδιά τους και να δημιουργηθεί μια κοινή ε, εμπειρία της οικογένειας, να υπάρχουν ευθύνες στην οικογένεια για την ανατροφή των παιδιών που θα μοιράζονται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και έτσι φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ευθύνη των γυναικών η ανατροφή των παιδιών. Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε η συμμετοχή των ανδρών ε, στην ε, οικογένεια και τώρα έχουμε περάσει και σε πιο λεπτά θέματα για την αξιοπρέπεια των γυναικών όπως το θέμα που αναφέρατε για την πορνεία και τη βιομηχανία του σεξ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η γενικότερη τάση των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τις επιβιώσασες, δηλαδή για τις γυναίκες ε, στο σύστημα της πορνείας, αλλά μιλάμε και για το θέμα της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή δεν θα υπήρχε πορνεία χωρίς τη ζήτηση, χωρίς τους άνδρες που είναι οι αγοραστές όπως είπατε. και που εκμεταλλεύονται την, ε, το ευάλωτο των γυναικών ε, και τη μη ισότητα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εξωθούνται οι γυναίκες και στην φτώχεια. Στην Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, βλέπω διαφημίσεις Οι γυναίκες, ξέρετε, στην πορνεία πρέπει να κάνουν τους άνδρες να αισθάνονται ότι οι γυναίκες στο σύστημα της πορνείας ε, πεινούν για σεξ και πρέπει να κάνουν τους άνδρες να αισθάνονται πρίγκιπες και επιθυμητοί. Και όλη η βιομηχανία του σεξ και η πορνογραφία αυτό το αποτέλεσμα προσπαθεί να επιτύχει στους άνδρες. και βλέπω αγγελίες που λένε ότι είμαι γυναίκα πεινασμένη για στοματικό έρωτα και κάθομαι στο αναπηρικό μου καροτσάκι ε, σε μια πολυκατοικία στα περίχωρα της Βουδαπέστης και περιμένω μόνο εσένα. Βλέπω λοιπόν μια τέτοια αγγελία και διαρωτώ με τι στρέβλωση υπάρχει στη σεξουαλικότητα και στην ηθικότητα των ανδρών. Και πόσο σημαντικό θα ήταν και οι άντρες να καταλάβουν πόσο τρελή είναι αυτή η κατάσταση. Και όλα τα προβλήματα ε, του συστήματος της πορνείας να τα κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι η δική τους η σεξουαλικότητα και η δική τους ικανότητα να έχουν μια υγιή και ευτυχισμένη σχέση με μια γυναίκα ε, είναι στρεβλωμένη. Και ε, αυτό το σύστημα της πορνείας, αυτός ο θεσμός της πορνείας υπονομεύει ακριβώς αυτά, αυτή τους τη δυνατότητα. Και ξέρουμε ότι από τα μέσα ενημέρωσης γνωρίζουμε ότι και οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές χρησιμοποιούν το σύστημα της πορνείας. Γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιείται και αυτός μέσω στην εκστρατεία σας κατά της πορνείας. Για την Ουγγαρία νομίζω κάποια παρανόηση υπάρχει, γιατί στο νέο σύστημα της Ουγγαρίας, στο νέο σύνταγμα της Ουγγαρίας δεν αναφέρεται καθόλου ότι είναι ε, παράνομη η άμβλωση. Νομίζω θα έπρεπε να αρχίσουμε να μιλάμε για το πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε άμβλωση, γιατί δεν είναι καλό πράγμα η άμβλωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή ε, η παράλογη ιδέα ότι η άμβλωση είναι καλό πράγμα. Η άμβλωση και ψυχολογικά και σωματικά ε, και ψυχικά είναι επιβλαβής για τις γυναίκες. Και εμείς, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των γυναικών, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε τις γυναίκες ώστε να αποφεύγουν τις αμβλώσεις. Και είναι πραγματική τραγωδία το ότι στον 21ο αιώνα τόσες πολλές γυναίκες χρειάζονται την άμβλωση που είναι τόσο τρομερό πράγμα. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τις ευθύνες των ανδρών για τον οικογενειακό προγραμματισμό και για την αντισύλληψη. Γιατί δεν είναι μόνο η υπευθυνότητα των γυναικών. Και πραγματικά ε, ε, έχω βαρεθεί τους άνδρες που λένε ότι είναι φεμινιστές και παλεύουν υπέρ του δικαιώματος των γυναικών για την άμβλωση αντί να σκέφτονται τα δικά τους, τις δικές τους ευθύνες στο να εμποδίσουν το να μείνουν οι γυναίκες έγκυοι χωρίς τη θέλησή τους. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ και ξαναδείτε το Ουγγρικό Σύνταγμα γιατί δεν θέτει την άμβλωση εκτός νόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ άλλοι τρεις ομιλητές και θα δώσω μετά το λόγο στην κυρία για να απαντήσει. κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω είναι από αυτές που είχαν την ιδέα να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών και που το οργανώσανε ε, όπως είναι δηλαδή με συνεργασία εθνικών οργανισμών, ευρωπαϊκών και εγώ δούλεψα, ήμουν αντιπρόσωπος από τη χώρα μου πρόσωπος και θα έλεγα ότι σήμερα το ευρωπαϊκό λόμπι ε, των γυναικών δεν το αναγνωρίζω έτσι όπως το φανταστήκαμε εμείς διότι εδώ και χρόνια βλέπω ότι αυτό που δημιουργήσαμε κυρίως για να συνοδεύσει την πολιτική για την ισότητα και των ευκαιριών για τις γυναίκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση φυσικά ένα οπλοστάσιο ε, οδηγιών σήμερα δεν ακούω κουβέντα για όλα αυτά και θα πρέπει να σας πω ότι αυτά που άκουσα σήμερα εκ μέρου τη εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Λόπου Γυναικών είναι κάτι το οποίο ιδεολογικά ε, με απογοητεύει βλέπω μια πτυχή προσέγγιση της αριστεράς χωρίς ε, ανοχή πολλοί έχουν αποκλειστεί. Μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε και με εθνικούς οργανισμούς που είναι πολύ ε, αντιπροσωπευτικοί. διότι πολλές προτάσεις από εθνικές οργανώσεις Φερπίν της Μάλτας δεν τις ταιριάζανε. Ε, με απογοητεύσαν λοιπόν διότι εγώ ήμουν πάντοτε Ε, με ενδιαφέρει πολύ η ευρωπαϊκή οργάνωση, αλλά δεν συμφωνώ ε, με το λόμπι, διότι αποφασίσανε Φερρυπίν ότι μια γυναίκα γίνεται ευρωβουλευτής Φερρυπίν, δεν έχει το δικαίωμα, αποκλείεται από τη συμμετοχή στα όργανα αυτού του λόμπι. Καταπληκτικό. Έπρεπε να το πω αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι είναι σοβαρό αυτό που βλέπουμε. Διότι τι βλέπουμε. Αποχή της ανοχής που το βλέπουμε συχνά και τις ε, ε, όλες τις κατηγορίες που ακούγονται από θρησκευτικές ε, ομάδες και την ανισότητα όσον αφορά τη σεξουαλικότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Εγώ να σας πω. Ε, εγώ να σας πω, εντάξει, συμφωνώ, ε, ανισότητα σεξουαλική ανάμεσα σε άντρες γυναίκες με ικανοποιεί, μα έτσι είναι. Είμαστε διαφορετικοί. Και εδώ δεν μπορούμε να πούμε με κατηγορίες. Τώρα, για την υγεία, τη σεξουαλική και της αναπαραγωγής, εγώ θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το λόμπι του ευρωπαϊκού λόμπι γυναικών δεν ακούμε για όλα αυτά, όλο για την πορνεία ακούμε. Εμείς έχουμε κάνει εκθέσεις όσον αφορά την πορνεία. Ξέρουμε περί μας πρόκειται. Εγώ έχω ψηφίσει τόσες και τόσες, να, ένα κάρο εκθέσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν, αν κατηγορείτε όταν κάνετε κατηγορίες σε σχέση με τη σεξουαλικότητα για τις γυναίκες, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει και μια ευθύνη των γυναικών. Δεν, μπορεί να δεν επιβάλλει κανείς στις γυναίκες πώς θα αντιθούν, πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα παρουσιάσουν το σώμα τους ή όχι. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η πτυχή. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πρόβλημα με αντικειμενικότητα. Λυπάμαι ειλικρινά όταν βλέπω τα νέα κορίτσια που παρουσιάζονται όπως, κάνουν, όπως το κάνουν σήμερα. Τι να κάνουν, δικαίωμά του είναι, επιλογή τους είναι, δίνονται όπως θέλουν. Θα, τις λέω λοιπόν συχνά, αν οι άντρες τις βλέπουν έτσι, τι γίνεται, δημιουργούνται ιδέες, ξυπνάνε επιθυμίες. Δεν εννοώ φυσικά ότι αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τι βιάσουν, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τι σημαίνει όμως και μια συγκεκριμένη πρόκληση. Για τι προκλήσει υπάρχει ευθύνη. Ευτυχώ στην εποχή μου δεν τα είχαμε, δεν είχαμε τα μέσα και μια χαρά ήταν τα πράγματα. Η αξιοπρέπεια μετράει. Λοιπόν, εγώ απογοητεύομαι αν ήξερα τι θα γινόταν τελικά αυτό το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, δεν θα ήμουν από αυτές που θα είχαν συμβάλει στη δημιουργία του. Ε, ε, Επόμενος, κύριε Σταραμπέλα. Κύριε, θα ήθελα να είσαστε σύντομος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να παραμείνουμε σε σοβαρό επίπεδο. Σχέση με τι δύο προηγούμενε παρεμβάσει, η κυρία Τάκεμπομ θα είναι ευτυχή και ο βελγικό μικρόκοσμο θα ε, γνωρίζει ότι πρόκειται για μια πρόσωπη τη άκρα ε, αριστερά. Ήταν ε, και βουλευτή τη φιλελεύθερη ομάδα στο Βέλγιο. Δεν είναι στο αριστερό τμήμα, αλλά είναι στο κέντρο δεξιό. Αυτή είναι η πολιτική γεωγραφία τώρα. Το θέμα της αυτοδιάθεσης των γυναικών, ε, δικαίωμα στην αντισύλληψη και στην ε, αμβλώσεις, κάτι το οποίο, για το οποίο ήμουν εγώ εισηγητής το 2010, ήταν η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που δεχόταν κατέβει το Κοινοβούλιο, αλλά δεν πυροβολούμε κάποια θρησκευτικά κινήματα, αλλά δεν μπορούμε να καταδικάζουμε το ενάμπλωση για να λέμε ότι είναι ένα έγκλημα και ταυτόχρονα να παρετούμε από τις αντισυλληπτικές μεθόδους και να ε, ε, ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντισύλληψη. Ξέρουμε, μοριστούμε στον 21ο αιώνα και υπάρχουν κάποιες ευθύνε. Ε, δεν ήθελα να πω αυτά τα πράγματα, διότι το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έχει άλλε δραστηριότητε από το να ασχολείται αποκλειστικά με την ε, σεξουαλική πτυχή, με το θέμα της βίας. Ε, φυσικά είναι σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Είναι μια γάγκρενα που αφορά όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κάνει διάφορους αγώνες ε, με επιτυχή αποτελέσματα όπως στην Ισπανία, αλλά αυτό αφορά και το, το κόσμο συνολό του. Πρόκειται για συνθήκες ειρήνης ή εμπόλεμες. Τώρα θα ήθελα να επικεντρώσω στην οικονομική πτυχή. Και για να συνεχίσουμε σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Σορτιέ για την πρόσβαση σε κάποιες εργασίες, να πω πόσο δύσκολο είναι το έργο σας, διότι τα μέσα έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά το φάσμα του πεδίου δραστηριοτήτων όλο και διευρύνεται. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο έχει προκύψει μετά την κρίση, ότι η, οικονομίες, οι χρηματοοικονομικές, χρηματοτραπεζικές, ε, εκεί που μας έχουν οδηγήσει και εκεί είδαμε όπου οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις και εκεί όπου οι γυναίκες είχαν θέσεις ευθύνης, είχαν ε, πειραστεί λιγότερο από την κρίση από ό,τι άλλους κλάδους. Ε, μιλάω για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, διότι ξέρουμε τι σημαίνει κρίση. Εξαφανίζονται οι γυναίκες. Ναι, όντως είμαστε διαφορετικοί, όχι μόνο φυσική και σωματική σκοπιά. το τονίσατε πολύ καλά κύριε, κύριε αλλά και για την αντίληψη των προγραμμάτων και το, και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη είχε πει ότι όταν <clears throat> ε, δανείζουμε μια γυναίκα, μας δίνεται μια αντιστάθμιση, ενώ αν δανείσουμε κάποιον άνδρα, κάποιον άνδρα όχι. Τώρα, σε ό,τι φορά την αγώνα εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλό επίπεδο ευθύνη, όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, εμεί δίνουμε το παράδειγμα στι χώρε μα, διότι σήμερα, ακόμα και αν δεν υπάρχει ισότητα, υπάρχουν 35% γυναικών εκλεγμένε στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν χώρε που έχουν πετύχει την ισότητα. Στην Ιταλία το 1 τρίτο των ε, της κυβέρνησης αποτελείται από γυναίκες, το 50% της κυβέρνησης αποτελείται από γυναίκες κλπ. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπου αυτή μπορεί να γίνει, υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να υπερβούμε την κρίση και διότι ο συμπεριφορά τον ε, συμπεριφορά αν επένδυνε γυναίκες τέτοιο στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι διαφορετική. Έχετε λοιπόν κάποια ε, θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα σύντομες παρεμβάσεις παρακαλώ. Κύριε Παπαδοπούλου και κύριε κυρία Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι παρακολουθώ τη δράση του Ευρωπαϊκού ε, Λόπι Γυναικών εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ήμουν παλαιότερα και στο Συμβουλίο της Ευρώπης και τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την αίσθηση και θα καταθέσω τη δική μου μαρτυρία ότι από τις πλήστες συζητήσεις που κάνουμε και σε αυτήν την Επιτροπή και αλλού σε σώματα που συζητούμε την ισότητα σε μεγάλο βαθμό αναλύσκουμε τους εαυτούς μας στο να μιλούμε όντως για τη γυναίκα θύμα για τη γυναίκα που είναι θύμα πορνείας, εμπορίας, βιασμών και αφήνουμε λίγο ε, πιο μακριά τη γυναίκα που μπορεί να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, ιδίως σε εποχές κρίσης. Με την οικονομική κρίση έχουμε δει ότι όντω και συμφωνώ με τις εκτιμήσεις σας υπάρχει οπισθοχώρηση όσον αφορά τις πολιτικές και για συμφιλίωση της οικογενειακής επαγγελματικής ζωής και για πρόθεση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπάρχει αύξηση της ανεργίας και όλα αυτά που έχετε πει. Να μην τα επαναλάβω, συμφωνώ απολύτω. Πέραν όμως από τη διάγνωση, Ειλικρινά ρωτούμε στο διατάφτα τι, τι ιδέων γενέστε, πώς λειτουργούμε ώστε να αξιοποιήσουμε την οικονομική κρίση ως μία πρόκληση και μία ευκαιρία. Του χρόνου θα έχει ευρωεκλογές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας και εδώ το Ευρωπαϊκό Λόπι Γυναικών μπορεί πραγματικά να κάνει εκστρατείε ενημέρωσης των γυναικών, να συμμετέχουν στις εκλογές και να αναδείξουν γυναίκες και άντρες που να είναι ευαίσθητες στα θέματα ισότητας. Τι παρεμβάσεις κάνουν το Ευρωπαϊκό Λόπι Γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στο Eurogroup. Πόσες γυναίκες υπάρχουν. Όταν αποφασίζουν, π.χ. για τη δική μας περίπτωση της Κύπρου, να προχωρήσουν σε κούρεμα ε, καταθέσεων αντί σε κούρεμα χρέου που έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ρίχνουν ουσιαστικά με τις αποφάσεις τους ένα λαό στη φτώχεια, τις γυναίκες και τη νέα γενιά στην ανεργία. Και ειλικρινά δεν ρωτούμε αν υπήρχαν εκεί γυναίκες που νιώθουν ότι όλες αυτές οι λαθασμένες αποφάσεις πραγματικά έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις και θα ρίξουν στην ανεργία νέες γυναίκες επιστήμονες με δύο-τρία μεταπτυχιακά. Θα ρίξουν μια γενιά κυρίως γυναίκες από φύτους με πολύ ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα να παραμείνουν ανεκμετάλλευτες ανθρώπινες εφεδρίες. Θα έπαιρναν αυτοί τα groups, το Eurogroup, η Τρόικα, τέτοιε αποφάσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ώρα που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε μεγάλα και παχιά λόγια και πρέπει να δούμε με ποιου συγκεκριμένου τρόπου μπορούμε να ενδυναμώσουμε μια άλλη σκοπιά των γυναικών, όχι τη γυναίκα θύματο, αλλά τη γυναίκα που πρωταγωνιστεί στι πολιτικέ αποφάσει, στι δράσει, στι κινητοποιήσεις που κατεβαίνει στους δρόμους και αντιστέκεται σε λαθασμένες επιλογές των τεχνοκρατών των Βρυξελών και η ερώτηση μου σε εσά συγκεκριμένα είναι αν διαθέτετε συγκεκριμένα στοιχεία ποια είναι η κατάσταση στις γυναίκες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που σήμερα πέραν από τις παραδοσιακές ανισότητες και τα στερεότυπα που αντιμετώπιζαν στις πατριαρχικές κοινωνίες πολλών χωρών Τούτη τη στιγμή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, πιθανόν αύριο στην Ιταλία, στη Σλοβενία και αλλού, πραγματικά αντιμετωπίζουν τρομερά οικονομικά προβλήματα και έναν πισωγύρισμα. Και δίνουν και την πρόφαση αυτέ οι οικονομικέ συγκυρίε στου εργοδότε να μην εργοδοτούν γυναίκε. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ε, ε, Λόμπι Γυναικών, να στηρίξει γυναικεία κινήματα σε αυτές τις χώρες και να ενισχύσει την παρουσία της γυναίκας. Ευχαριστώ. Děkuji, pane předsedo. Já nechci mluvit dlouho a děkuji za vaši zhovývavost. Ehm, Já bych chtěla podčarknout, paní, co řekla paní Teitelbaum o prostituci. There is no translation in English. Δυστυχώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία προς το παρόν τουλάχιστον. Alors, je, je vais essayer de le dire. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γαλλικά, ίσως να είναι πιο εύκολο. Η κυρία Μπάουν ε, μίλησε για πάρα πολλά ζητήματα, θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ όλη την μέρα για να τα αναλύουμε. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που μου είπε σχετικά με την ε, πορνεία. Είπατε ότι η Επιτροπή μας ε, έχει εγκρίνει πολλές και ποικίλε εκθέσεις για την βία, αλλά Κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων δέκα ετών υπήρξαν τρεις εκθέσεις που δεν ενέκρινε η Επιτροπή μας. Ήταν η έκθεση ε, για τη βιομηχανία του σεξ, για την ε, πορνεία και τι επιπτώσει στην ε, υγεία και την ακαιρεότητα των γυναικών, αλλά και στην σεξουαλοποίηση των, των κοριτσιών. Νομίζω ότι πρόκειται για θέματα ιδεολογικά και πολιτικά τα οποία μας εμπόδισαν να υπερσυφίσουμε αυτές τις τρεις εκθέσεις, διότι αυτές τις τρεις εκθέσεις είχαν εγκριθεί. Τα είχαμε πάει ακόμη πιο μακριά. Θα σα ευχαριστήσω πάλι στο Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών για την εκστρατεία τους επί της ε, πορνείας. Ήμουν παρούσα όταν ε, έγινε η παρουσίαση αυτή της αυτής σημαντικής πρωτοβουλίας. Πραγματικά η πρωτοβουλία Not for Sale δεν είναι προσπόληση δηλαδή. Ήταν μια εκστρατεία πολύ πετυχημένη όπου εξήγησαν το όλο γεγονός ε, και είπαν ότι δεν είναι μόνο ε, οι γυναίκες που πέφτουν θύματα, αλλά είναι και το όλο σύστημα που προκαλεί αυτή την κατάσταση. Και θα πρέπει λοιπόν να απορρίψουμε την ε, πορνεία στο συνολό της και όχι την καταναγκαστική πορνεία. Ευχαριστώ. Θα σας ε, ε, υποδείξω ως μοντέλο σύντομης παρέμβασης. Ευχαριστώ. Δυστυχώς έχουμε λίγο χρόνο στη διδασή μας κυρία Τέτερμπαουμ, θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας μετά από όλες τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά για να υπάρχει τουλάχιστον ισότητα γλωσσική, αφού πριν μίλησα αγγλικά. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί κανείς να νιώθει ότι απογοητεύεται από μια οργάνωση, αλλά νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έχει ως στόχο το να είναι μια προοδευτική δύναμη, αλλά όχι εξτρεμιστική πάνω σε μια πολιτική σκακέρα. Για μας είναι σημαντικό να δίνουμε, προβλήματα, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των γυναικών σήμερα. Είναι πολλά τα προβλήματα αυτά. Είχα μόνο ένα τέταρτο για να μιλήσω, επομένω δεν μπορούσα πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ. Υπάρχει όμως ε, και η σελίδα μας, στην οποία μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές μας, για να ολοκληρωθεί λοιπόν η σημερινή μου επίσκεψη, σας παρακινώ να δείτε την ιστοσελίδα μας με όλα τα σχετικά στοιχεία. Θα δείτε και πολλά στοιχεία για τις πρωτοβουλίες μας και μπορώ να σας ενημερώνω κι εγώ. Όταν ε, μιλάμε για τις γυναίκες, πολύ συχνά προσπαθούμε να μετατοπίσουμε τις ευθύνες, είτε για να πούμε ότι οι γυναίκες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, είτε για να λέμε ότι οι άνδρες πρέπει να αναλάβουν ε, την ευθύνη αντί των γυναικών. Νομίζω ε, ότι η αρχή του θέματος ισότητας ανδρών και γυναικών είναι αυτή η, ο σωστός καταμερισμό ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία και δεν θέλουμε να μειώσουμε τις ευθύνες των μεν και να αυξήσουμε τις ευθύνε των δε. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομη και θέλω να πω ότι δεν λαμβάνονται αποφάσεις που να βασίζονται σε ηθικές αξίες είτε αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση γιατί έχετε δίκιο εσείς που είπατε ότι είναι τρομερό πράγμα η άμβλωση κανείς δεν θέλει να ευχηθεί σε μια γυναίκα την άμβλωση η συζήτηση όμως αλλού τίθεται όταν έχουν ακολουθηθεί όλες ε, οι εναλλακτικέ λύσεις ή όταν δεν δόθηκε η δυνατότητα να ακολουθηθούν όλες οι εναλλακτικέ λύσεις, εμείς που θέλουμε να έχουν πλήρη επιλογή οι γυναίκες, θέλουμε να έχουν επιλογή για το σώμα τους. Περί αυτού πρόκειται. Δεν λέμε ότι η άμβλωση είναι καλή λύση, γιατί καμία γυναίκα δεν πρόκειται να πει θέλω να πάω να κάνω άμβλωση. Δεν τίθεται έτσι η συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να αφορά τα δικαιώματα των γυναικών να διαθέτουν το σώμα τους όπως θεωρούν σκόπιμο και δεν θα κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση σε σχέση με αυτό. Το ε, να υπάρχει στην Α ή στη Β χώρα μια τέτοια συζήτηση, στην Ουγγαρία παραδείγματο χάρη μια τέτοια συζήτηση, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μετατοπίζει ε, το βασικό θέμα σε σχέση με τις αξίες τις οποίες υπερασπιζόμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη θα πρέπει να είναι μόνο θετική εξέλιξη. Συχνά παρουσιάζονται οι γυναίκες ως θύματα, όπως είπατε, και πρέπει να βρεθούν κάποια πρότυπα, να βρεθούν κάποια πρόσωπα που να προωθούν την εικόνα της γυναίκας και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για ένα τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι που εμείς οι γυναίκες πρέπει συστηματικά να το συμπεριλαμβάνουμε στις απαντήσεις μας, να δίνουμε μια θετική εικόνα της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας και να κερδίζουμε όσον αφορά την προσέγγιση μας σε αυτό το οποίο επιδιώκουμε και αυτό το οποίο προσδοκούμε από την κοινωνία. Και είναι κομμάτι του αγώνα των γυναικών αυτό. Και στον τρόπο παρουσίαση των πραγμάτων ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής επ' αυτού και ίσως επ' αυτού να έχετε δίκιο. Σε σχέση με τις ηθικές αξίες, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο η άμβλωση το συζητήσιμο θέμα. Σε σχέση με την πορνεία, η θέση μας δεν βασίζεται σε ηθικά κριτήρια. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και οι γυναίκες που λαμβάνουν το λόγο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών δεν ε, κάνουν μια ηθική αξιολόγηση. Οι αξίες της ισότητας ανδρών και γυναικών, το προβαλλόμενο μοντέλο, η εικόνα των γυναικών και οι ζημίες επί της υγείας, αυτά είναι τα κριτήρια. Δεν είναι, τα κριτήρια δεν είναι το τι θέλει να κάνει οποιοδήποτε στη ζωή του. Ούτε θέμα ε, πίστης ή απιστίας έναντι του συντρόφου. Δεν τίθεται με ηθικούς όρους η συζήτηση. Είναι μια συζήτηση επί των αξιών. Και ε, εκεί πρέπει να παραμείνει η συζήτηση. Όσον αφορά τη θρησκεία, ανέφερα πολλά κριτήρια πολιτικά, οικονομικά, ανέφερα και τα θρησκευτικά κριτήρια εδώ και χρόνια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών ε, συμμετέχω ε, σε σχετικές συζητήσεις για το καθεστώς των γυναικών και είτε προέρχεται από το Βατικανό, είτε από το Ιράν, είτε από την Αίγυπτο, είτε από οποιαδήποτε χώρα, το ότι η θρησκεία προβάλλεται ως πρόφαση για να δικαιολογηθούν πράξεις βίας κατά των γυναικών ή πράξεις ε, που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις ως Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και στο πλαίσιο της ισότητας ανδρών και γυναικών δεν μπορούμε παρά να τα καταγγείλουμε όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να αποκρύψουμε ένα από αυτά τα θέματα που αποτελούν τμήμα των συνολικών προβλημάτων. Και τέλος, όσον αφορά την οικονομική πτυχή, όντως δεν το ανέφερα εν εκτάσεις στην παρέμβασή μου, γιατί δεν είχα χρόνο να περάσω σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά έχετε δίκιο ότι Σήμερα οι γυναίκες δεν είναι τα μόνα θύματα, αλλά συχνά είναι τα πρώτα θύματα ή τα κύρια θέματα των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται όσον αφορά την οικονομική κρίση και έχετε απολύτω δίκιο επ' αυτού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δράσεις τις οποίες εμείς διεξάγουμε σχετικά και στην πρώτη μας διεθνή ε, ε, Γενική Συνέλευση στο Ζάγκρεπ ε, θα αναφερθούμε και στα οικονομικά προβλήματα. Το είχαμε αναφέρει και πέρυσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Όμως είμαστε ένα λόμπι, ασκούμε πίεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ υπάρχει και η δυσκολία στο να είναι κανείς μέλος ενός ε, εκτελεστικού οργάνου ευρωπαϊκού και να έχει και ε, θέση εδώ, γιατί εδώ ασκούμε μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε ε, να ε, τονίσουμε το ρόλο των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και για τις επερχόμενες εκλογές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ένα πρόβλημα mentoring με γυναίκες ευρωβουλευτές που συνοδεύουν ε, νεότερες γυναίκες ε, με υπόβαθρο μετανάστευσης για να υποστηρίξουν αυτές τις γυναίκες που έχουν ακόμη λιγότερο ευκαιρία πρόσβασης. 35% των βουλευτών είναι γυναίκες και μόνο 2% έχουν υπόβαθρο μετανάστευσης. Επομένως το ποσοστό αυτών των γυναικών είναι ακόμη μικρότερο και γι' αυτό προσπαθούμε να δράσουμε ακριβώς εκεί που είναι περισσότερο ευάλωτα τα πρόσωπα και όσον αφορά τις ποσοστώσεις ε, κάνουμε σχετική δουλειά και όσον αφορά ε, την συμμετοχή των γυναικών στην ε, λήψη αποφάσεων στον οικονομικό τομέα και στην καταπολέμηση όλων αυτών των μηχανισμών που φύγουν διπλά τις γυναίκες και στις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και στη μερική απασχόληση και στη διαφορά μισθολογικών αποδοχών πολύ συχνά οι γυναίκες ε, θίγονται πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Και στις συντάξεις ε, επίσης υπάρχει επίπτωση για άλλη μια φορά. Είναι λοιπόν θέματα προτεραιότητας ε, στον αγώνα που κάνουμε καθημερινά και κάνουμε και πολλές δημοσιεύσεις και δουλεύουμε με σχετικά Ινστιτούτα και δείκτες Βλέπω όμως ότι ο πρόεδρος ε, με κοιτάζει επίμονα γιατί θέλει να κλείσω την παρέμβασή μου. Στην ιστοσελίδα μας λοιπόν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να σας αναφέρω σήμερα. Συμφωνώ πάντως μαζί σας όσον αφορά την ένδυα των γυναικών και δυστυχώς σήμερα οι γυναίκες είναι ακόμη περισσότερο θύματα της κρίσης από ότι οι Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο. Σαφώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και θέλουμε να το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο και γι' αυτό αφαιρώνουμε και πολύ χρόνο. Είμαι πεπισμένο ότι θα υποφεληθούμε από τις γνώσεις σας και από την εμπειρία σας ε, σε σχετικά θέματα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε στην Επιτροπή μας και που είχατε αυτή τη συνάντηση μαζί μας. Also, we, we have, we have... Κοιτάξτε. Έχουμε 15 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την πρωινή συνεδρίαση. Μία πρόταση. Να αναγγείλω πως ε, το λόμπι των ε, γυναικών για την Ευρώπη έχει ε, οριστεί ως οργάνωση για το Νόμπελ και αυτό νομίζω θα πρέπει να το δηλώσουμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. <clears throat> Πρόκειται για την ε, φιλοκτονία. Έχουμε πρόβλημα διότι δεν υπάρχει χρόνος ε, και έχω ε, και έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Χάζα Ζαϊνάμπ Μπαγκούρα αλλά προηγούμενα θα πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση περί φιλοκτονίας. Η κυρία Παδοπούλ θα λάβει το λόγο και λυπάμαι που δεν θα έχουμε χρόνο για να το εξετάσουμε σαν πάνω στο ζήτημα. Έχετε το χρόνο. Το λόγο κύριε Παδοπούλ. Chair, I will try to be very brief. Θα φροντίσω να είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Προετοίμασαμε μια έκθεση για την φιλοκτονία, είναι μια έκθεση πρωτοβουλία. Μιλάω για φιλοκτονία, ο ορισμό είναι σαφή. Πρόκειται για ένα ουδέτερο ε, όρο που αφορά την ε, μαζική ε, θανάτωση προσώπων ή εμβρίων, είτε είναι ασθενικά είτε γυναικεία, δεν γιατί είδαμε από το 1990 Εκατό εκατομμύρια γυναίκες θεωρούνται ότι έχουν εξαφανιστεί και υπάρχουν κολλήσει που ξεκολουθούν με φύστα τι πρώτε διακρίσει όσον αφορά τον προκαθορισμό του φίλου του βρέφου, τι αυλώσει για εγκατάλειψη ή τη ανάπτυξη τη ηλαιών βρεφών μυστικά και μόνο λόγω του φίλου. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Και ο βασικό λόγο είναι κάποιε ε, ιδέε και κάποιε προκαταλήψει ε, που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές του κόσμου και οφείλονται σε πολλούς λόγους σε κάποιες ε, κοινωνίες ε, θεωρείται ότι οι... τα κορίτσια δεν προσφέρουν πολλά στην ε, οικογενειακή ζωή και στο οικογενειακό εισόδημα και αυτές οι πρακτικές δυστυχώς συνεχίζονται. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ε, προτιμούν τα αγόρια από τα κορίτσια και αυτές οι αντιλήψεις ε, εντείνονται και με ιδιαίτερε περιοχές που δεν υπάρχουν κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια. Στόχος αυτής της έκθεσης ε, είναι να καταπολεμηθεί η φιλοκτονία αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά όλες τις όλες τις προκαταλήψεις ε, που οδηγούν σε παρόμοιες καταστάσεις και να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση των ε, πληθυσμών για αυτές τις πρακτικές, ε, να δείξουμε όλες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η συνειδητοποίηση και οι διακρίσεις που υφίστανται το γυναικείο φύλλο και να μπορέσουν να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές, να υπάρξουν χρηματοδότηση και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων των Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα κράτη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πολιτικό διάλογο και να ενισχύσουμε τις εθνικές νομοθεσίες προκειμένου να αποφευχθεί η φιλοκτονία, να προλάβουμε το κοινωνικό περιβάλλον και το πολιτιστικό, να βελτιώσουμε την πρόσβαση της γυναικών στην ιατρική περίθλιψη, στα μικροδάνεια και μηχανισμούς για τις οικογένειες και τις γυναίκες και να αποφεύγονται κάποιες επιλεκτικές ε, επιλογές στον τομέα του φύλου. Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλία και ενθαρρύνουμε και τους υπόλοιπους βουλευτές να προωθήσουν ιδέες μέσω τροπολογιών όταν αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλία θα ε, κυκλοφορήσει στις διάφορες γλώσσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω να λάβει το λόγο η κυρία για Μπρόσκα, διότι είναι συνδυσμένε σύντομε παρεμβάσει, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ, είστε σύντομοι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι αληθινό πολιτικό θέμα και το βλέπω αυτό στην έκθεση πρωτοβουλία και συγχαίρω την κυρία Παπαδοπούλου. Όντω το 2008 και εγώ ήμουν δραστηριοποιημένη ε, ήμουνα στη θέση του Πρόεδρου μας και ζήτησα να γίνει μια ακρόαση εδώ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Λίκον Τζον ε, είναι σε ένα παγκόσμιο δίκτυο για τα δικαιώματα των γυναικών και ασχολείται πάρα πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών και δει στην Κίνα ε, όπου έχουμε και την πολιτική όπου κανεί, μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα παιδί. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα Πρώτον, για τον ορισμό. Αυτή η έκθεση ε, αφιερώνεται στις γυναίκες όπου αντιμετωπίζουν διάφορα ε, προβλήματα και όλα αυτά με βάση με το φίλο τους. Εκπλήσωμε που δεν κοιτάξαμε δεν ε, τονίζεται η πλευρά που έχει να κάνει με την ε, τυχή της γυναίκας σε σχέση κυρίως όταν μιλάμε για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ε, εκτρώσεις. Ορισμένοι όροι δεν είναι κατάλληλοι για μένα, δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του θέματος. Δηλαδή όταν κάποιοι όροι μου δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τη μετάφρασή του σε κάποιε άλλε γλώσσε, ή στη δικιά μου, στα συλλογικά, στα γερμανικά. Θα ήθελα να δούμε μήπως μπορούμε να δούμε από κοντά τα θέματα των μεταφράσεων να υπάρχει σωστή αποδόση. Όταν αφορά το φύλλο και αυτό που λέμε gender και sex υπάρχει συχνά διαφορετικός τρόπος μετάφρασής τους. σε σχέση με τη γυναικεία φύση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο καμιά φορά να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο gender και φύλλο. Σεξ. Ε, να μην δούμε μόνο το θέμα της ε, να δούμε το θέμα που έχει να κάνει ε, όχι μόνο κάποια θέματα που έχουν όχι με την μη παρουσία της γυναίκας αλλά τις συνέπειες που έχουν ε, στα παιδιά σε σχέση με τα παιδιά και την απουσία της μητέρας, να δούμε όλα αυτά, να δούμε τις στατιστικές, διότι υπάρχουν όντως στατιστικές όσον αφορά αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα έχω και πολλά άλλα να πω, αλλά δεν θέλω να καταστρατηγήσω το χρόνο που μας είπατε ότι είναι λίγος κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο προς συζήτηση. Νομίζω ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά στην έκθεση αυτή και ε, υπάρχει καλή ισορροπία σε αυτά τα οποία επικρίνονται και τονίζεται παράλληλα και η σημασία του να έχουν οι γυναίκες ε, το δικαίωμα της ακεραιότητας στο σώμα τους. Νομίζω ότι θα κλείσουμε όμως εδώ τη συζήτηση. Η προθεσμία και τις τροπολογίες είναι οι 3 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΦΑΜ 19 Ιουνίου. Και θα πρέπει τώρα να σταματήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα ε, διότι έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να καλωσορίσουμε εδώ την κυρία Μπαγκούρα, που είναι ειδική εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε περίπτωση σειράξεων. Έχει οριστεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μουν. ήταν παλαιότερα υπουργό στη Σιέρα Λεόνε και έχετε 20 χρόνια εμπειρίας στα θέματα της διπλωματίας σε πολιτικά και σε πρακτικά ζητήματα. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα σας δώσω τον λόγο για να κάνετε μια παρέμβαση και θα συζητήσουμε αργότερα, θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, γιατί δεν έχουμε το χρόνο για συζήτηση τώρα. Ξέρω ότι έχει λήξει ο χρόνος και ζητώ από τους διερμηνείς να μείνουν ε, λίγο περισσότερο. Ε, το τελευταίο τμήμα της ε, συζήτησης θα γίνει μόνο στα αγγλικά. Λοιπόν, έχετε το λόγο για να μην καθυστερώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα στην Επιτροπή σας για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ηθικό ζήτημα της εποχής μας το να σταματήσει η σεξουαλική βία σε περιπτώσει σειράξεων. Είναι πρώτη μου επίσκεψη στις Βρυξέλλες ως ειδική εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών και με τιμά το ότι λαμβάνω το λόγο σε αυτή την επιφανή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη μου επίσκεψη. Η σεξουαλική βία που έχει σχέση με το φύλλο είναι έγκλημα από μόνο του. Από την αρχαιότητα θεωρεί το αποδεκτό ε, οι στρατιώτες σε περιπτώσεις πολέμου να βιάζουν ε, γυναίκες και κορίτσια και ε, αυτό ήταν ένα τρόπος, ένας τρόπος υποβάθμισης του εχθρού. Η διεθνής κοινότητα δεν κατάφερε να θέσει τέλος στις σειράξεις, όμως επιτέλους αναγνωρίστηκε η ιδέα να αντιμετωπιστεί η βία σε περιπτώσεις πολέμου και οι τραγικές συνέπειες που έχει αυτό στην ακαιρεότητα των προσώπων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ιστορικές πρωτοβουλίες για την εξάλληψη αυτών των εγκλημάτων. Από το 2010 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει θεσπίσει ψηφίσματα χωρίς προηγούμενο που αναγνωρίζουν το εύρος αυτού του προβλήματος και που δίνει ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση του προβλήματος. Τα ψηφίσματα αυτά 18 18-28 και 19-60 και το 2025 αποτελούν το πλαίσιο και για τη δική μου δουλειά ως ειδική εκπροσώπου καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας της σειράξης. Το ψήφισμα του 2000 ζητεί από τα κράτη παγκοσμίω να αναγνωρίσουν αυτό το πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα και να σταματήσει η ατιμορρησία για τα σεξουαλικά εγκλήματα και αυτό να είναι κάτι το οποίο θα ενταχθεί σε όλες τις προσπάθειες ειρήνευσης το ψήφισμα επίσης ζητεί από όλα τα συμβαλόμενα μέρη και από όλους τους συμμετέχοντες σε πολέμους να προστατεύσουν γυναίκες και κορίτσια από τη σεξουαλική βία και από τους βιασμούς κατά τη διάρκεια των σειράξεων. Το ψήφισμα 18-20 ήταν το πρώτο ψήφισμα των ΗΠΑ που αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως τακτική πολέμου και θέμα διεθνούς πολιτικής ε, σχετικά με την διατήρηση της ειρήνης. Το ψήφισμα 1888 βασίζεται στα προηγούμενα ψηφίσματα, το 2025 και το 1820 και δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν μέτρα διεθνώς ε, και ζητείται από την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων να προσθέσουν κριτήρια σε σχέση με τους βιασμούς και άλλες πράξεις σεξουαλικής βίας. Το ψήφισμα 1888 επίσης ε, ζητεί τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που η δουλειά τους ε, θα υποστηρίζει τους εθνικούς μηχανισμούς απόδοσης δικαιοσύνης, ώστε να ε, εφαρμοστεί πλήρως το ψήφισμα 18-20. Τέλος, το ψήφισμα 19-60 ζητάει να δημιουργηθεί ένα βήμα και ένα μηχανισμό παρακολούθησης και ανάλυσης για ε, να έχουμε καλύτερη γνώση αυτών των εγκλημάτων και να γνωρίζουμε καλύτερα ε, πότε διαπράττονται τέτοια εγκλήματα σε περιπτώσεις πολέμου. Αυτά τα ψηφίσματα μα έχουν δώσει το διεθνές νομικό πλαίσιο και του μηχανισμού παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, ε, ούτω ώστε να μπορούμε να καταγγείλουμε και να καταδιώξουμε τους δράστες. Για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι βασικέ αιτίε αυτών των ε, συγκρούσεων ούτως ώστε να εξαλείψουμε αυτές τις περιπτώσεις ε, βίας. Στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις σειράξεις τονίζεται το ότι επιδίωξη των στοιχείων πλούτου που είναι αιτία πολέμου αποτελεί αιτία και για την σεξουαλική βία. Στην ε, δημοκρατία του Κογκό χρησιμοποιήθηκε ο ε, βιασμός ε, ε, ως μέσο παρεμπόδισης των μονάδων του πληθυσμού που προσπαθούσαν να εμποδίσουν την καταλήστευση των, του ορυκτού πλούτου. Και στην Κολομβία επίσης χρησιμοποιήθηκε η σεξουαλική βία σε περιπτώσεις που προσπάθησαν να εμποδίσουν την καταλήστευση του εθνικού πλούτου. Η εξόριξη ορυκτού πλούτου έχει άμεση σχέση με τη διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων και οι ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν ότι στο Ανατολικό Κονγκό συνεχίζουν οι εμπλεκόμενοι στις σειράξεις να εποφελούνται ε, από τον ε, έλεγχο των ορυχείων για την εξόριξη χρυσού ε, και άλλων ευγενών μετάλλων από το εμπόριο αυτών των ε, ορυκτών ε, που έχουν ε, τεράστια αξία τροφοδοτούνται οι σειράξεις και η σεξουαλική βία. Υπάρχουν σπάνιες γέες που χρησιμοποιούνται για τα κινητά τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες που είναι αντικείμενο που οδηγεί σε αυτές τις σειράξεις. Οι συνθήκες στα ορυχεία είναι πάρα πολύ σκληρές. Η καταναγκαστική εργασία χρησιμοποιείται και πολλές φορές τα παιδιά είναι αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και χρησιμοποιούνται και στα ορυχεία και είναι και θύματα σεξουαλικής βίας ο πλούτος ε, θα έπρεπε ε, να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων και όχι να τροφοδοτεί τον πόλεμο λόγω της ε, επιζήτησης του ορυκτού πλούτου. Μπορούμε να εξαλείψουμε αυτές τις αιτίες πολέμου, δηλαδή την επιδίωξη του ορυκτού πλούτου. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ζητούν από τις... το ψήφισμα 1887 ζητά από ε, τις χώρες να λάβουν μέτρα ε, κατά της ε, εξόριξης ορυκτού πλούτου που οδηγεί σε καταλήστευση και σε σεξουαλικά εγκλήματα. Δεν θα πρέπει να υποφελούνται ένοπλες ομάδες από την προσπάθεια εξόριξης ορυκτού πλούτου. θα πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε την ε, σωστή διαχείριση και την ορθή διακυβέρνηση στη δημοκρατία του Κογκό καταπολεμώντας τις πράξεις των ομάδων που επωφελμιούν τον ορυκτό πλούτο και καταλήγουν σε σειράξεις. Εάν εξασφαλιστεί ε, η εξάλληψη της δουλείας και της σεξουαλικής βίας που έχουν άμεση σχέση με την εξόριξη του ρηκτού πλούτου, τότε πραγματικά θα έχουμε επιτύχει κάτι. Είναι μία από τις βασικές αιτίες των σειράξεων η επιζήτηση ορυκτού πλούτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα σημαντικό μερίδιο στο διεθνές εμπόριο αυτών των ε, πρώτων υλών και επομένως παίζουν και σημαντικό ρόλο όσον αφορά αυτές τις σειράξεις. Η σχετική νομοθεσία ε, θα θέσει τα κατάλληλα πρότυπα για, τις, ε, την εξόριξη ορυκτού πλούτου στον Ανατολικό Κογκό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε προσφάτως ότι θα θέσει 3 εκατομμύρια ευρώ για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας και άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ για την εκπαίδευση των τοπικών φορέων, για την οικονομική συνεργασία και για την ε, για την εκπόνηση δραστηριοτήτων και οδηγιών για τη δέουσα επιμέλεια. Πρέπει να ακολουθήσετε ισχυρή γλώσσα όταν επιβάλλετε την, υποβάλλετε την έκθεσή σας στο πλαίσιο ε, του ε, δημοσίου διαλόγου, ούτως ώστε να είναι ισχυρά τα νομοθετικά μέτρα που θα ληφθούν. Η πραγματική νομοθεσία, η σκληρή νομοθεσία για τα θέματα της εξόριξης μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα και στη δημοκρατία του Κονγκό και αλλού. Θα πρέπει ο ρηκτός πλούτος να μην συνεισφέρει στην βία, αλλά να, αποτελέσει, να αποτελέσει ένα καταλήτη για την ευημερία του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. thank you. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά το ότι ήρθατε και μας επισκεφθήκατε, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και τώρα θα θέλαμε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις μεταξύ σας. Δυστυχώς δεν θα συμβεί εδώ, αλλά και τώρα, αλλά σε μισή ώρα σε ένα, μια άλλη αίθουσα. WIB 4 4 στην αίθουσα Βίλι Μπραντ, στον τέταρτο όροφο, στο αίθουσα 4. Στη 1 και 10 θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 2 και εκεί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να έχουμε ανταλλαγή απόψε μαζί σας. Ευχαριστώ.